Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής ΙΝΤΑ στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι όλοι θα έχετε την ημερήσια διάταξη. Θέλετε καμία αλλαγή, από ό,τι φαίνεται όχι. Οπότε θα προχωρήσουμε. Σημείο 2, οι ανακοινώσει του Προέδρου. Συνομιλία χωρίς μικρόφωνο μέσα στην αίθουσα. clear and για, για κάποιο λόγο έχει αλλάξει το μικρόφωνο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να μιλάτε αργά, καθαρά και με σαφήνεια. Οπότε, προχωράμε απευθείας στην πρώτη ψηφοφορία επί του σημαντικού αυτού νομοθετήματος τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία, θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, ώστε να διαπιστώσουμε Ναι, ναι, θα το κάνουμε αργά-αργά, αφού μου το ρωτάτε. Λοιπόν, να βρούμε τις κάρτες της ψηφοφορίας. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Πάρτε όλοι τις κάρτες σας, παρακαλώ. Μάρτι, γνωρίζεις εδώ πώς λειτουργεί η συσκευή ψηφοφορίας. Λοιπόν, αρχίζουμε τη δοκιμή. Δεν λειτουργεί. Πέρα Okay, and the test Πέρας της δοκιμαστικής ψηφοφορίας δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα είναι εντάξει και με τα θέματα των πολιτικών ομάδων. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Έλεγχος ξένων άμεσων επενδύσεων, ξένων επενδύσεων. 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν. Τροπολογία. 2, 0, 1. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν, χωριστή ψηφοφορία επί της τροπολογίας 27. Το πρώτο μέρος της 27 Καταπίπτη, το δεύτερο μέρος του πρώτου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατόπιν, συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4-1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4-2 υπέρ. Κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 27 από την άφετη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 27 δεν ήταν τσίτρε. 27 ήταν από την Άφετ. Oh, ναι. 27 της άφετα απορρίφθηκε. Και κατόπιν. Συμβιβαστική 4-3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2-9-6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 303 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν στο 338 το δεύτερο μέρος υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «370 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τρία το δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. εννέα ένα. υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 της άφετ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9-2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9-3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και έχουμε δύο ταυτόσιμες τροπολογίες, η 4.15 και 4.16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η συμβιβαστική 9-5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική 5α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν έχουμε τη συμβιβαστική 9, 5 β. Είναι, ναι. Συμβιβαστική 9, το μέρος 5 ε, β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9, μέρος 5 γάμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 54 από την, της Ήτρε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κατόπιν, συμβιβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και την συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 68. Έλεγχος για την 68. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα οι σκεψεις σκέψεις. Συμβιβαστική R1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. R2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ, 81. Ήρεμα και συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική R3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R, R5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά Ήτρε, τροπολογία 4, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, παραλείψαμε την 97. Παραλείψαμε την τροπολογία 97. Υπέρ της 97. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική R8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R10α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και κατόπιν η 9 της ΕΚΟΝ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική R12α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R12β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R12C υπέρ κατά αποχές. νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε. R12C έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας σαφώς εγκρίνεται. Υποθέτω ότι κάτι θα άλλαξε εντωμεταξύ. Συμβιβαστική R13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R15α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R16α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R20α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική R 21α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα το παράρτημα συμβιβαστική άνεξ 1α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική άνεξ 1β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία η επόμενη καταπίπτει, καταπίπτει, καταπίπτει και μετά έχουμε μία ψηφοφορία, η τελευταία ψηφοφορία, έναρξη ηλεκτρονικά Λοιπόν, τελική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, τον κύριο Προύστ. Εγκρίνεται με σημαντική πλειοψηφία. So, now I Προύστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους κοιόδης εισηγητές που συνεισέφεραν για αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Στην τελευταία μας συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών είπα ξεκάθαρα το εξή. Θέλω την υποστήριξή σας για να ξεκινήσω διαπραγματεύσεις με βάση τις ε, ε, τροπολογίες με βάση το άρθρο 69C, όχι, όχι να αποφύγουμε τη συζήτηση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, όντως, αλλά γιατί δυστυχώς το χρονοδιάγραμμα δεν είναι προς ωφελός μας. Ξέρετε πολύ καλά τι προθεσμίες έχουμε και επειδή υπάρχουν και οι προθεσμίες για τη μετάφραση, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναβληθεί θεωρητικά για τον Ιούλιο η ψηφοφορία. Οι τριμερείς διάλογοι μπορούν να ξεκινήσουν μόνο το Σεπτέμβριο επομένω και η Επίτροπος μου το επιβεβαίωσε και τις προάλλες και μπροστά σας ότι το Συμβούλιο προχωράει από τη δική του μεριά στις συζητήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν κρίμα νομίζω να περιμένει το Συμβούλιο την απόφαση του Κοινοβουλίου, ενώ έχουμε καλές συμβιβαστικέ τροπολογίες που την υποστηρίζουν ε, πολύ. Η Βουλγαρική Προεδρία, την οποία συνάντησα, έκανε πολλή προσπάθεια και αυτό το κείμενο θεωρείται προτεραιότητά της, επομένως μπορούμε να αποφύγουμε να χάσουμε δύο μήνες, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο για τη θητεία μπροστά μας. Σας κάνω λοιπόν την εξή πρόταση. Αυτό το κείμενο που όπως ξέρετε ε, το περιμένουν οι επιχειρήσεις μας, και πολλές επιχειρήσεις ο χρόνος είναι θέμα αποτελεσματικότητας, ρεαλισμού, επομένως λογικό θα ήταν να κερδίσουμε αντί να χάσουμε αυτούς τους δύο μήνες. Σας προτείνω βεβαίως να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση με βάση τις ε, τροπολογίες που υπερψηφίσαμε στην Επιτροπή Ίντα. Αυτά δύο λόγια ήθελα να σας πω και ξανά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Προύστ. Υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ των τροπολογιών στην Επιτροπή Ίντα και λόγω των χρονικών περιορισμών ο εισηγητής ζητάει με βάση το άρθρο 69C να ξεκινήσουμε διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ζητάει την εντολή σας εδώ για, να, για την ψηφοφορία. Οι διαπραγματεύσεις, η διαπραγματευτική ομάδα έχουμε τον πρόεδρο της ΣΥΝΤΑ, τον σκιώδη εισηγητή και, τους, ε, και τον εισηγητή. Συμπεριλαμβάνεται και ο κ. Μπουτικόφερο, εισηγητής της ΙΤΡΕ επίσης και οι διαπραγματεύσεις μπορούν ε, να ξεκινήσουν αφού αναγγελθεί η απόφαση στην Ολομέλεια στις 11 Ιουνίου. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Για αυτό που ζητάει ο εισηγητής, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το αίτημα του εισηγητή, για να του δοθεί εντολή δηλαδή. Ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, πήραμε την, πήρε την εντολή. Θα το αναγγείλουμε λοιπόν στην Ολομέλεια και μετά θα ξεκινήσει πάρα αυτά η διαπραγματευτική ομάδα της διαπραγματεύσεως. Σας ευχαριστώ για την ξεκάθαρη ε, πλειοψηφία. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα προς ψηφοφορία. Συνδέεται με το πρώτο, φαντάζομαι. Είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας έκθεση του κυρίου Winkler. Με πολλές τροπολογίες. Κοίταξα προσεκτικά τις τροπολογίες. Μην ξεχνάτε ότι σύμφωνα ε, με το άρθρο 54 πρέπει να ε, συνεργαστούμε με την ΑΦΕΤ. Και λόγω των, του ιστορικού που υπάρχει ανάμεσα σε εμά και στην ΑΦΕΤ θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά τις ε, τροπολογίες αυτές της ΑΦΕΤ. Καμία από τις επιτροπές δεν θα αμφισβητήσει τις αρμοδιότητες και τα προνόμια της άλλης από τις συζητήσει που είχα. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 46 είναι μη παραδεκτό. Γιατί αφορούν τις αρμοδιότητες της ΑΦΕΤ. Η Γκουε θα ήθελε να πει ότι δεν θα συμμετάσχει στον συμβιβασμό 3B και το συμβασμό 4B. Μετά λοιπόν από αυτέ τι ανακοινώσει ξεκινάμε την ψηφοφορία. Η πρώτη είναι ο συμβιβασμό ένα. Πέπ. Κατά. Αποχέ. Διοθετείται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 11 που θα είναι μια προσθήκη στο συμβασμό του προηγούμενου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 3α υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 3b υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 4α υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 4β υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 40. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 41 είναι συμβατός, συμβατή μάλλον με την τροπολογία, με την ε, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Εν συνεχεία, έχουμε την τροπολογία 46. Μόνο στο πρώτο τμήμα θα ψηφίσουμε τώρα, γιατί το δεύτερο τμήμα είναι μη παραδεκτό όπως σας είπα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, τη 46, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. αποχές, Υιοθετείται. Συμβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 79 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. υιοθετείται. Συμβαστική. Τύπος. 12. Ελέγχουμε την συμβαστική, όχι, την τροπολογία 86. Ψηφίζουμε τώρα της προφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 12 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Διοθετείται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά, αποχές υιοθετείται. 91 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές τη 13, τη συμβαστική τροπολογία 13 ψηφίζουμε τώρα. Συμβαστική Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 100 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 101 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 103 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 17, συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. 111 του κ. Βίνκλερ υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Και τώρα συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Με πολύ πλατιά πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Βίνκλερ. Εκτός μικροφώνου. Δεν είμαι σίγουρη για την 41 το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν ξέρω αν μπορούμε τέτοια ώρα μετά από τόση ώρα να το κάνουμε. 41. Κανονικά δεν μπορεί να γίνει έλεγχος ε, τόσο καθυστερημένα. Ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Απερίφθη αυτή η τροπολογία. Α, όχι, πέρασε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 41. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Ναι. 36 ψήφισαν και εγκρίθηκε. Είναι καλύτερα αν σηκώνατε πιο ξεκάθαρα τα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε τα διάφορα, το αγαπημένο μου θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. 20 Ιουνίου εδώ στις Βρυξέλλες, λέει ο Πρόεδρος, θα συνεδριάσουμε.